Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ που ήρθατε τόσο πρωί. Αλλά τι να κάνατε μου ψηφίζουμε. Έχουμε απαρτία και μπορούμε λοιπόν να αρχίσουμε Πρώτο σημεία στην ημερησία διάταξη. Ειδικά μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη-μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Στις 16 Φεβρουαρίου ανταλλάξαμε απόψη σε ενέκτακτη συνεδρίαση και αποφασίσαμε βάσει του άρθρου 15.2 του κανονισμού να προχωρήσουμε σε απλουστευμένη διαδικασία με τροπολογίες. Μετά από διαβουλεύσεις με τους συντονιστές, η πρόεδρος συνέταξε σχέδιο έκθεσης για συγχρηματοδότηση μέχρι και 100% για να υποστηριχθούν οι δράσεις ε, σε, επαντώντας σε φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Λιγότερο το 5% θα πρέπει να αφορά αυτό ε, στα κράτη-μέλη για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η προθεσμία για αντιρρήσεις από το 1 δέκατο των μελών της Επιτροπής έληξε στις 17 Μαρτίου το απόγευμα. Δεν ε, έλαβε η Πρόεδρος ε, ούτε η Γραμματεία καμία αντίρρηση μέχρι την εκπροή, οπότε θεωρείται εγκεκριμένη η έκθεση. Άρα, προτείνω να ζητήσουμε η βάση του άρθρου 69C ε, εντολή από την Ολομέλεια για την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων με μία και μοναδική τροπολογία προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση που εγκρίθηκε. Η διαπραγματευτική ομάδα, η πρόεδρος και η συγγήτρια και οι σκιώδεις συγγητές. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ αυτά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε. And the decision is... Εγκρίνεται η απόφαση κατά πλειοψηφία. This is unique. Thank you. Thank you very much. This... Ευχαριστώ πολύ. Uh, Δεύτερη ψηφοφορία. Έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Νοβάκοφ. Ο σωστό συνδυασμό χρηματοδότηση για τι περιφέρειε τη Ευρώπη, εξορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρετε την ιστορία τη έκθεση, είχαμε συζητήσει. Κύριε Νοβάκοφ, θέλετε να πείτε τίποτα. Uh, we go straight to... Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Και σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε. Η τροπολογία 24 ψηφί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 25 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 26 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 30 είπε. κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Μάλιστα. Την 30 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία. Φέρες. Απορρίπτεται. Σας ευχαριστώ. Η τροπολογία 31. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές. Για να το αυτό. Παρακαλώ τη 42 ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. The vote is closed and Απορρίπτεται. Α, τώρα έχω καταλάβει το ταμπλό. Η 43 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα πάμε στη συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Ψηφί κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα θα πάμε στις ε, προτάσεις της Επιτροπής Προπολογισμού 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται. η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί η τροπολογία 89 επέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η, η τροπολογία 94 επέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, έχουμε τις προτάσεις του προϋπολογισμού 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προτάσεις της μετυπής προεπιλογισμού παρθμόνου. 9 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί αλλά στην μου. Την 9 έτσι το προπολογισμό αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. The vote is closed. Απορρίπτεται. Οι προτάσεις της Επιτροπής Προπολογισμών, παρθμών 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 149 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τσεκ καλά ελέγχουμε λοιπόν την 157 ηλεκτρονικά αρχής δόρυψη η λήξης. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 17 ψηφίπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 171 ψηφίπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ. Ωραία. Ας το ελέγξουμε. Την 171 ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 172. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προτάσεις προπολογισμού περιθμών 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προτάσεις Επιτροπής Προπολογισμού Υπαριθμών 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τώρα έχουμε προτάσεις από την Επιτροπή Γεωργίας. A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκριση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκριντή, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι ή ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι F υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι H υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγρι άι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα έχουμε αριθμούς άγκρι 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άγκρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές Απορρίψετε. Άγκρι 11 υπέρ κατά αποχές Απορρίψετε. Άγκρι 12 υπέρ κατά αποχές Απορρίψετε. άκρη Do we... Oh, 12. Tell me. 13. Uh, 13. Άγκρι... Πάμε στη 13. Τη Επιτροπή Γεωργία. Μα είναι τόσε πολλές, δεν τα χάνει κανεί. Είπε. No, it's uh, a little bit more. Ε, ε, ε, λίγες έχουν μείνει. Δεν γίνεται unblock. Υπάρχει μία στη μέση που δεν μπορεί να ψηφιστεί μέση. 13 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 23 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρη 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκρή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Νοβάκοφ μου. Here we go. And we continue now Thank you. with our next... Uh... να επόμενη εκθέση συντάκτρια είναι η κυρία Κρεσό. Παράτηση τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για τον Λογοταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Δεν είναι παρούσα η κυρία Μπρέσο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν λοιπόν με την ψηφοφορία. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην προφορική τροπολογία επί της 81. Υπάρχει κάποιος που να είναι κατά όχι, άρα θέτω σε ψηφοφορία την 81 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπάρχει ε, ένσταση στην προφορική τροπολογία όχι. 83 με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80, ε, συγγνώμη, συμβιβαστική 2. Κατα, ε, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 103 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά 8, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχουμε 126 Υπάρχει ένσταση στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφορία την 126 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 139 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. 14, συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Α ελέγξουμε την 14, γιατί δεν είμαι και σίγουρη. 14, γιατί 14 ψηφίζαμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι τροπολογία 14. Ψηφίστε παρακαλώ. Λογικά θα δουλεύει το σύστημά σα Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρα και εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε στην 21 προφορική τροπολογία. Υπάρχει ένσταση. Όχι. Ψηφορία επί της 21 με, με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 έχει καταπέσει, καταπίπτει. Γίνουμε στην αιτιολογική σκέψη 6. Με προφορική τροπολογία δεν υπάρχει ένσταση, λοιπόν. Ε, τροπολογία για το 6 με την... Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ συμβαστική Εγκρίνεται. Η συμβαστική 17. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ε, με την προφορική τροπολογία δεν υπάρχει ένσταση. Ψηφίζουμε για αυτήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά προχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε. Αλλά ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 66. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην, στην αιτιολογική σκέψη 21. Υπάρχει προφορική τροπολογία, υπάρχει ένσταση. Όχι, επομένω ψηφίζουμε γιατί είναι 21 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση, όπως τροποποιήθηκε. Ευχαριστώ. Okay. The next, the next uh, vote will be on the assessment of Horizon 2020 implementation. Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 2020 με γνώμονα την ενδιάμεση αξιολόγησή της και την πρόταση για το ένατο πρόγραμμα Πιλέσιο. Θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Φαν Μίλτενμπουργκ. Όχι, ωραία. Προχωράμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται, συγγνώμη. 25. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ Υπέρ κατά αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται. Αποχές. Α, συγγνώμη, δεν είδα καλά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ψηφίζουμε για το τελικό κείμενο. The vote Έγκρινεται λοιπόν η ε, γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κύριε Φαν Μιλτενμπεργκ. Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Έχουμε την ε, δυνατότητα σύνδεσης ίντερνετ ε, για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή η Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Gigabyte και του 5G. Κύριε Λιούερ, έχετε να πείτε κάτι. Ναι. Κοιτάξτε, συνήθως ε, δίνουμε τις ε, εκθέσεις του συναδέλφου, αλλά αποφάσισα αυτή να την αναλάβω εγώ ε, και ξέρω πως δεν ήθιστε, αλλά τώρα γνωρίζοντας, μάλλον ήθιστε να ευχαριστούμε τους συναδέλφους ε, για τη συνεργασία και για την εξέβρεση καλών συμβιβαστικών. Ε, το λέω πραγματικά. Υπέρ λοιπόν της πρώτης συμβαστικής ή κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. And uh, our last vote for today. Uh, Τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα λοιπόν είναι αυτή που αφορά την εισήγηση της κυρίας Νταμάτο, προαγωγή της σύνδεσης στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Νταμάτο μου? Όχι. Ε, ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με την ε, ψηφοφορία για τη συμβαστική. Ένα υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64, 65 με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές, 67 συγγνώμη, ναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβι, ε, συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές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 το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά. Άρχεται. The vote is closed. And... Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ πολύ. So, uh, in this point... Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες και τελειώνει η ώρα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλά δουλέψαμε. And, uh, our, our next, uh, Επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. I ask you to keep silence. Λίγη ησυχία παρακαλώ. If anybody is leaving the room, do it. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ ησύχως ή δυνατόν. Possible. No. Μάλλον δυνατόν Okay, we continue now with the consideration of the draft. Συνεχίζουμε. Έχουμε το σχέδιο έκθεσης κυρίας Βέστφαλ με τον ενδιαφέροντα τίτλο «Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020». Στα τέλη του περασμένου έτους αποφασίσαμε να κάνουμε σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ένωσης μετά το 2020 με τον τίτλο που σας ανέγνωσα. Και ορίσαμε συγγήτρια την κυρία Βέστφαλ. Η έκθεση αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει την πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα βασικά χαρακτηριστικά του εξυγχρονισμού της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 εν ώψη και των μεταρρυθμίσεων που έχουν προβλεφθεί για τον Ιούνιο του 2017. Κάναμε ένα εργαστήριο για τα δομικά στοιχεία αυτά, έτσι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με το Policy Department Β τον Ιανουάριο, το τμήμα μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα θα ψηφίσουμε σε έκτακτη συνεδρίαση το Μάιο. και Προτείνω ε, να ορίσουμε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών την 30η Μαρτίου. Θα έχετε αρκετό χρόνο μέχρι τότε για να συνεδριάσουν και οι και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Βέστφαλ για να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καταρχάς σε όλους, ακόμα και αν πέρασαν ήδη οι ε, ψηφοφορίες, ε, πραγματικά κυρία Πρόεδρε δεν είναι μόνο ενδιαφέρον ο τίτλος αλλά και η δουλειά ολόκληρη για την έκθεση αυτή και αυτή που μας περιμένει για τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής έχει ήδη αρχίσει. Τι εννοώ. Δεν εννοώ μόνο το ερώτημα για το ποιες μεταρρυθμίσεις έχουν νόημα ή τι βελτιώσεις χρειαζόμαστε. Εχθές είχαμε εδώ τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, και καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ε, μετά το 2020 υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική ε, συνοχής, η περιφερειακή. Ακούμε ε, τι λέει ο κύριος Γιούνκερ και το σενάριο 4 στην πρότασή του και σιγά σιγά αρχίζω να αμφιβάλλω εάν και κατά πόσο υπάρχει τέτοιο μέλλον. Μετά διάβασα και μια συνέντευξη της Επιτρόπου κυρίας Γιούροβα και με ζώσαν τα φίδια ε, σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, διότι λέει ρητά ότι δεν ξέρει πάρα πολύ καλά, δεν ξέρει ακριβώς πόσα χρήματα θα υπάρξουν στο μέλλον για την πολιτική συνοχής και παραθέτω, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν καν κονδύλια για την πολιτική συνοχή. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή μην καταργηθεί η πολιτική συνοχή. Αυτό το καταπληκτικό μεγαλειώδη εργαλείο ευρωπαϊκής Αλληλεγγύη, Αυτό το μοναδικό μέσο ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία, Αυτό το εργαλείο που κάνει την Ευρώπη απτή, χειροπιαστή, επιτόπου στα μάτια των πολιτών δεν επιτρέπεται να καταστραφεί. Αυτό το τονίζει και η έκθεσή μου και το ξεκαθαρίζει πολλαπλώς. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ισχυρή πολιτική συνοχής και σύγχρονη. Ε, αλλά εδώ ισχύει και κάτι άλλο. Ορισμένα πράγματα πρέπει να παραμείνουν όπως έχουν και άλλα να βελτιωθούν. Καταρχά θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι θα μπορούσε να παραμείνει ως έχει. Πιστεύω ότι είναι εκ των όνου κάνευ υπαρκής χρηματοδότηση. Η περιφερειακή πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί ε, στα καθήκοντά της όταν έχει περισσότερα χρήματα, όχι λιγότερα. Εκτός αυτού, η γενική δομή της περιφερειακής πολιτικής έχει νόημα και είχε νόημα και πρέπει να διατηρηθεί. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, να ενισχύονται όλες οι περιφέρειες στην Ευρώπη. Και εδώ θέλω να επιμείνω. Βεβαίως να έχουμε το κέντρο βάρους στις λιγότερο ανεπτυγμένες, αλλά και οι λεγόμενες μεταβατικές και οι πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες χρειάζονται ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζονται ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό έχει πετύχει από κάθε άποψη. Και τη θεματική συγκέντρωση τη θεωρώ σημαντική να φύγουμε από την αρχή ε, που λέει δίνουμε λίγα χρήματα σε όλους, σαν το ποτιστήρι που ποτίζουμε αδιακρίτως, ε, και να επικεντρωθούμε σε εκείνα τα έργα που προστατεύουν το περιβάλλον, που έχουν ανάπτυξη και που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Τώρα έρχομαι, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτά που ε, χωράνε βελτιώσει. Τα εξή τρία. Πρώτον, και δεν είναι και κανένα μυστικό αυτό, η απλούστευση. Το συζητάμε συνέχεια. Αυτό το θέμα μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Όλο και περισσότερο βλέπουμε παράπονα και καταγγελίες για υπερβολική γραφειοκρατία. Θα πρέπει αυτό το γραφειοκρατικό άχθος να μειωθεί. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ιδιαίτερα είναι να σπάσει ένας φαύλος κύκλος. Εκείνοι ε, που υποβάλλουν τις αιτήσει κάνουν λάθη και μετά βγαίνουν νέοι κανόνες για να αποφεύγονται αυτά τα λάθη. Οι νέοι κανόνες όμως κατά κανόνα οδηγούν σε ανασφάλεια και αβεβαιότητα οπότε νέα λάθη. Άρα γιατί να μην ακολουθήσουμε τελείως διαφορετικό δρόμο και μη συμβατικό αν θέλετε. Τι εννοώ. Όποιος ε, όλα αυτά τα χρόνια έχει υποβάλει αιτήσει χωρίς λάθη και χωρίς πρόβλημα. Ίσως θα πρέπει να ελέγχεται σπανιότερα και να έχει πιο απλές διαδικασίες. Κοινή κανονισμένη για όλα τα ταμεία και αυτό το ακούμε πάντα. Είναι το δεύτερο ε, και αυτό θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη δουλειά επιτόπου. Από τις συνομιλίες που είχα γνωρίζω επίσης ότι η εναρμόνιση ε, των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Εκτός αυτού θα μπορούσα να φανταστώ πάρα πολύ καλά μια τράπεζα δεδομένων για τις ενισχύσεις αυτές, ένα είδος πλατφόρμας ή μια, ένας κόμβος στο διαδίκτυο που να μπορούν με μια ματιά οι δήμοι και οι κοινότητες να ενημερώνονται. Επόμενο θέμα, η ε, ευελιξία. Μ' αρέσει αυτή η θεματική συγκέντρωση. Ταυτόχρονα όμω, θα πρέπει οι Δήμοι και οι περιφέρειές μας να είναι σε θέση να αντιδρούν σε απρόοπτα. Ας πούμε, κρίση του προσφυγικού παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ας πούμε, τεχνική πρόοδος και τεχνολογική σε κάποιες περιφέρειες. Εκεί θα πρέπει να μπορούν να αντιδρούν Δήμοι και περιφέρειες. Για να υπάρχει λοιπόν αυτή η ευελιξία, τι προτείνω ένα κλάσμα των ε, πόρων από τη συνοχή, να το αφήνουμε στην άκρη και να βλέπουμε μετά από 4-5 χρόνια ποιες είναι οι νέες προκλήσεις για να μπορούμε να διδρούμε γρήγορα. Θα θεωρούσα σωστό ας πούμε ένα τέτοιο αποθεματικό να δημιουργείται σε επίπεδο προγραμμάτων. Και από εκεί και πέρα θα ήταν καλό να είναι και τα επιχειρησιακά προγράμματα προσαρμοσμένα και να μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και έρχομαι στο τρίτο τώρα. Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ και πάρα πολύ σκληρά και επιτύχαμε να υπάρχει αρχή της εταιρικής σχέσης. Πρέπει να ενισχυθεί. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε κάποιες περιφέρειες λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτό, σε κάποιες άλλες λιγότερο καλά και σε κάποιες καθόλου. Άρα θα μπορούσα να φανταστώ πάρα πολύ καλά για να διατηρηθεί αυτή η αρχή να ε, επιβάλλουμε μια υποχρέωση. Πολύ σύντομα μερικά ακόμα σημεία. Δεν θα σας εκπλήξει αυτό που ζητώ. τα αποτελέσματα της αστικής ατζέντα να μπουν και στην επόμενη ε, πραγματική περίοδο και να είναι πιο ορατά τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα υπάρξει χωριστή έκθεση, γι' αυτό το αναφέρω μόνο εμπαρόδο, αλλά πρέπει να το αναφέρω και στη δική μου έκθεση. Εκτός αυτού, ε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα χρηματοδοτικά μέσα ε, μπορούν να είναι χρήσιμη συμπλήρωση. Αλλά η περιφερειακή πολιτική ε, βασίζεται κυρίως σε επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Ποια είναι τώρα τα πεδία πολιτικής ή τομής πολιτικής ακόμα και αν δεν υπάρχει διάδοχη στρατηγική από τη στρατηγική του 2020, κατά την άποψή μου τα διαρθωτικά ταμεία θα πρέπει να φροντίζουν για νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ε, καινοτομία και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω δύο λόγια για τη διαδικασία. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να έχει τελειώσει μέσα Ιουνίου εγκαίρω για το Φόρουμ Συνοχής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε το Μάιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία που θα έχουμε με τους κοιόδης ηγητέ. Και επίση χαίρομαι για τις ιδέες που σίγουρα θα συμπληρώσουν την έκθεση. Στο άρθρο 16 ε, πήρα κάποια στοιχεία ε, που πρότεινε ο Λάμπερτ Φανίστερ Ρόιτ και έχουμε συμφωνήσει διακομματικά. Ενδεχομένως μπορούμε να διαφωνούμε σε κάποια θέματα, όλα αυτά πιστεύω να μην είναι πάρα πολλά αυτά και να μην έχουμε ε, δεκάδες τροπολογίες ε, που να αποδυναμώσουν τελικά το κείμενο. Θα πρέπει να δώσουμε εμεί σκληρή μάχη για τη συνοχή ε, και η μάχη αυτή δεν θα πρέπει να δοθεί μεταξύ μας. Ο εχθρός είναι απέναντι ο μεγάλος αγώνας και η μεγάλη μάχη που θα δοθεί είναι να διατηρηθεί στο μέλλον ε, η πολιτική συνοχής και τα διορθωτικά ταμεία. Εγώ θέλω ε, να είναι αυτή απλή, ευέλικτη, στραμμένη προς το μέλλον, εύκολη στην εφαρμογή και με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Ποιο είναι ο στόχος μου. Να έχω μια έκθεση σαφή, σχετικά σύντομη, ε, ευανάγνωστη και ευνόητη έτσι ώστε να δώσουμε ε, στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο αυτόν τον αγώνα που σας λέω. Ευχαριστώ πολύ. now we will begin. Ευχαριστώ κύριε Βέσφαλ. Αρχίζει η συζήτηση με τους πιο συγγητές. Ο κύριος Χέτμαν είναι ο πρώτος. Thank you, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της αυτή. Είναι εξαιρετικό ανάγνωσμα. Και συμφωνώ και συνυπογράφω τα περισσότερα από όσα γράψατε εδώ. Βέβαια θα έχω και κάποια σχόλια, αλλά Πιστεύω πως η βάση για συμβιβασμό είναι πολύ στερεά κάποιο σχόλιο έχω να κάνω. Όταν συζητάμε την πολιτική συνοχή μετά το 2020, με λυπεί το γεγονός ότι πρέπει πάλι να πούμε πως είναι η πιο σημαντική πολιτική επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διατηρηθεί και να συνεχιστεί. Εάν αμφισβητείτε, νομίζω πως θα ήταν τεράστιο λάθος ε, για την Ένωση, όπου συχνά μιλάμε για προώθηση της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε αυτή η πολιτική να καταστεί πιο ορατή και μας εντυπωσιάζει που οι πολίτες πολύ συχνά δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, αλλά πραγματικά να ρωτιέμαι πώς ε, θα μείνει ικανοποιημένο ο κόσμος από αυτή την πολιτική αν εμείς οι ίδιοι και οι εσωτερικές μας συζητήσεις αμφισβητούν ε, την πολιτική αυτή και έχω την εντύπωση ότι οι ίδιοι πρέπει να πιστούμε μεταξύ μας ότι πρόκειται για την πιο σημαντική όντως πολιτική που έχει ποτέ ασκηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία όπως και η συγγήτρια ότι πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα μέσα για αυτή την πολιτική μετά το 2020 και το Brexit δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να περικοπεί ο προπολογισμό και για να επιβληθούν μέτρα ε, λιτότητας. Δεν μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία. Εάν λοιπόν θέλουμε αυτή η πολιτική συνοχής ε, να ε, ε, είναι αισιόδοξη και να προωθεί την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των πολιτών, τότε οφείλουμε να ε, μαζευτούμε, να ανασκουμποθούμε και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και αν αυτό το καταφέρουμε, δεν θα χρειάζεται πια η προώθηση της πολιτικής συνοχής. Επίσης, κάτι που είναι γνωστό σε όλους, απλοποίηση, το ανέφερε και η συγκεντρία. Οι δικαιούχοι της πολιτικής αυτής ε, συχνά ε, <clears throat> χάνουν την, την, την ε, ενέργειά τους γιατί τους την δαπανούν μέσα σε όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να φτάσουν στα χρήματα. Αν είχα ένα όνειρο λοιπόν, το όνειρο μου θα ήταν όλος αυτός ο κόσμος που, που συντάσσει τους κανόνες, τους όρους και τα κριτήρια ε, για την κάθε πολιτική, μια φορά να βρεθεί στην άλλη πλευρά του θρανίου, του, του τραπεζιού. Να προσπαθήσουν δηλαδή να συντάξουν ένα project, να το υποβάλουν ώστε να πάρουν χρήματα οι ίδιοι και μετά να υποστούν και τον έλεγχο που οι ίδιοι έχουν φτιάξει. Νομίζω πως πολλά θα άλλαζαν τότε. Τώρα, συνέργειες Δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω. Ε, πρέπει να υπάρχει συνέργεια ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα, ας πούμε, Horizon 2020, εύση ε, και αν πραγματικά υπάρχει σύνδεση και συνεργασία, τότε το αποτέλεσμα της πολιτικής συνοχής θα είναι επίσης πιο ορατό. Τρίτο σημείο, ευελιξία. Είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο και καλός προγραμματισμός για το τι και πού θα ε, δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα. Αλλά τη σήμερα ημέρα οι αλλαγές ε, στην πράξη είναι τέτοιο είδους ε, όπου πρέπει να ενταχθεί εδώ και κάποια ευελιξία. Γιατί διαφορετικά η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Πρέπει, οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι για να μπορούμε να ενσωματώσουμε τις ε, αλλαγές. Ε, τώρα, εταίροι, δεν χρειάζεται εδώ να μπω σε λεπτομέρειες γιατί η συγγήτρια τα ανέφερε όλα αυτά πολύ αναλυτικά. Οι επιδοτήσεις θα πρέπει να διατηρηθούν και άλλα μέσα να συμπληρώσουν τις ε, χορηγίες, τις επιδοτήσεις αυτές. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε τη δυνατότητα εισαγωγής μιας μειχτής, αξιολόγη, μιας μειχτής διαδικασίας, δηλαδή ε, να έχουμε τις επιδοτήσεις και ταυτόχρονα και δάνεια, για παράδειγμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν κάποιος δικαιούχος έχει καλά εφαρμόσει το πρόγραμμα, τότε, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να καταργούνται τα επιτόκια ή ένα κομμάτι του χρέους να διαγράφεται τεράστιο κίνητρο θα ήταν κάτι τέτοιο και ώστε να κάνουν και άλλοι δικαιούχοι ε, σωστά τα προγράμματα. Πιστεύω πως έτσι θα έχουμε όλα ένα και περισσότερους ε, δικαιούχους που θα υλοποιούν προγράμματα εάν προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και το πιο σημαντικό για μένα, ε, για να μπορέσουν όλα αυτά να πετύχουν και να λειτουργήσουν, έτσι ώστε όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ και οι βουλευτές μετά από μας να μην χρειάζεται ξανά μανά να συζητούν <clears throat> το γιατί αυτός ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Αυτές τις αλλαγές λοιπόν πρέπει τώρα να τις κάνουμε, ώστε όλα να λειτουργούν έγκαιρα, στην ώρα τους, να ξεκινούν όλα μαζί, εμείς λοιπόν πρέπει πρώτα να τελειοποιήσουμε το σύστημα και το πρόγραμμα. Ίσως να σας φανεί ότι προκαλώ, αλλά πιστεύω πως είναι κατάλληλη στιγμή όχι μόνο να δείξουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής, αλλά ίσως να πρέπει να δείξουμε και στους πολίτες ποια είναι η πραγματικότητα, ποια, μάλλον θα ήταν η πραγματικότητα γύρω τους εάν δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την πολιτική συνοχή θα μπορούσαμε να τους δείξουμε με πώς θα οι κοινότητες χωρίς τη βοήθεια της πολιτικής συνοχής. Να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι χωρίς αυτές τις δεκάδες χιλιάδες project πολύ λιγότερες θέσεις απασχόλησης θα υπήρχαν, πολύ λιγότεροι δρόμοι, λιγότερα έργα και πολύ χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Σα ευχαριστώ. ακούγοντα τον εισηγητή και την εισηγήτρια μάλλον και τον συνάδελφό μου έχω καλυφθεί ε, είπαν όλα όσα ήθελα να πω έκαναν όλες τις προτάσεις που θα ήθελα να κάνω και συμφωνώ πλήρως μαζί τους. Συμφωνώ κυρίως με τον προλαλήσαντα, τον συνάδελφο. Ε, βεβαίως, χρειάζεται να συνεχίσει η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Ε, κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Βεβαίως, χρειάζεται ευελιξία. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο που ανέφερε η κυρία Χέτμαν που είναι πολύ σημαντικό για την πολιτική ομάδα, το ECR, και είναι το ζήτημα των συνεργειών μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων αφενός και των διαρθρωτικών ταμείων αφετέρου. Νομίζω ότι αυτό, αυτή η συνεργεία, αυτή η συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των δύο ταμείων θα πρέπει να βελτιωθεί. Και θα ήθελα αυτό να ε, φαίνεται πιο ξεκάθαρα και στο τελικό κείμενο της ε, έκθεσης. Θα υποβάλουμε τροπολογίες που θα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. θα τονίσουμε την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει συνέχεια στην πολιτική συνοχή και να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή στο μέλλον. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασε η συγγήτρια ή ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοδομητική στάση και να υποστηρίξουμε την ε, έκθεση. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος όλοι θα συμφωνήσουμε και θα είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε uh, Ευχαριστώ. Μην Πριν αρχίσουμε να παίζουμε με τα τουβλάκια για το πώς θα χτίσουμε την επομένη πολιτική συνοχή, να δούμε πρώτα τα θεμέλια. Θα το κρεμίσουμε όλο το οικοδόμημα της πολιτικής συνοχής. Ε, θέλουμε να χτίσουμε κάτι ε, έτσι από θεμέλια ή έχουμε μια ε, αρκετά ε, μετριοπαθή ανακαίνιση. Μάλλον προς το δεύτερο το πάει η και συμφωνώ απολύτως. Όλο το πλαίσιο, το βασικό της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει να διατηρηθεί μετά το 2020. Υπάρχουν όμως βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν και από το ισχύον πλαίσιο. Ας πούμε, ισολογιστικό έλεγχο ή τους ελέγχους γενικά και συμφωνώ με τις προθέσεις της εισηγήτριας. Θα πρέπει πραγματικά να έχουμε ένα σύνολο κανόνων για όλα τα διαρθωτικά ταμεία και ένα ενιαίο σύστημα ελέγχων και πληροφόρηση. Για την ευελιξία επίσης συμφωνώ με τα μέτρα που προτείνει και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πρόταση του κανονισμού Omnibus. Χρειάζεται αυτή η ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το προσφυγικό π.χ. Άρα, συμφωνώ με την κυρία Βέστφαλ ότι χρειαζόμαστε ε, μία ε, εγκάρσια ε, πρόταση για να προετοιμάσουμε και το νομοθετικό πακέτο μετά το 2020. Πλην όμως υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης για την ευελιξία που έχω κάποια ερωτηματικά εγώ. Με, αυτό έχει να κάνει με την εξή ιδέα. Ότι θα πρέπει να έχουμε, λέτε, ένα αποθεματικό για απρόπτα γεγονότα, για πάνε ενδεχόμενο και τη δυνατότητα αναπρογραμματισμού. Όπως γνωρίζουμε, οι αναπρογραμματισμοί κονδυλίων γίνονται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις και θα πρέπει να είναι πολύ καλά ισορροπημένοι. Αυτό γενικά μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό και να υπονομεύει τη σταθερότητα και την ε, προβλεψιμότητα της πολιετούς στρατηγικής επενδύσεων. Διερωτώ λοιπόν αυτό το αποθεματικό πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ποια είναι αυτά τα πρόοπτα. Υποθέτω ότι θα πρέπει να συνδέεται με τους θεματικούς στόχους. Ε, αλλά θέλω να ακούσω τι γίνεται εάν ε, οι ε, περιφέρειες δεν χρησιμοποιήσουν, δεν απορροφήσουν αυτά τα χρήματα. Τι θα απογίνουν. Σύμφωνο με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Είμαι αναφανδόν υπέρ διότι ε, είναι ένα κίνητρο για υγιείς πολιτικές και δημοσιονομικές και οικονομικές. Επιπλέον ε, μειώνεται ε, η μη προβλέψιμη ε, δαπάνη. Εγώ είμαι και κατά της εδαφικής ε, διάστασης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αν θέλουμε να έχουμε καλύτερο οικονομικό συντονισμό και καλύτερη οικονομική στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να επιμείνουμε στην εστίαση ακριβώς και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, διότι έχει να κάνει με τις εθνικές μακροοικονομικές πολιτικές και αν αρχίζουμε να το βάζουμε αυτό σε ε, επίπεδο περιφερειακό θα χάσουμε και την ε, λογοδοσία του προγράμματος και το στόχο. Επίσης, κάτι άλλο που προτείνει η συγγήτρια έχει να κάνει με τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική αλλαγή. Είναι πραγματική πρόκληση και μπορούν να παίξουν ρόλο τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά όχι με απλή αύξηση των ε, πιστώσεων. Οι περιφέρειες που έχουν πρόβλημα δημογραφικό χρειάζονται ένα πολύ ευφύη τρόπο χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων. Για να μην έχουμε διαρροή εγκεφάλων θα πρέπει να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην περιφέρεια για να επενδύσουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό τελικά θα κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια. Και ένα τελευταίο διαπεριφερειακή συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό καλύπτεται από το Interreg Αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες που συνεργάζονται σε διάφορες πρωτοβουλίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Interreg και δεν μπορούν να επενδύσουν ε, παράδειγμα σε προγράμματα επίδειξης ε, ε, ε, των προϊόντων τους. Μόνο τα αλλαγή πληροφοριών μπορούν να έχουν από το ίντερεξι διασυνοριακά. Για να διευκολύνουμε λοιπόν τις επενδύσεις, θα πρέπει να αυξήσουμε ε, τον προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Συνεργασία, ταφική όπως λέγεται, και στα πλαίσια του τρέχοντος ε, προγράμματος Interreg για ε, άμεσες επενδύσεις στις περιφέρειες στο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιό της και ελπίζω μαζί με τους υπολείπους Κιώδης και την εισηγήτρια φυσικά να βελτιώσουμε την έκθεση και να γίνει ακόμα πιο φιλόδοξο εγχείρημα. Γιατί τελικά μας χρειάζεται και αυτή η φιλοδοξία για να προχωρήσουμε στην πολιτική συνοχή μετά το 2020. Ευχαριστώ. Και να τη συνεχίσουμε δηλαδή. Ευχαριστώ κυρία Νταμάτο. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Βέστο για αυτή την πρώτη έκθεση ε, που αφορά την ε, πολιτική συνοχής μετά το 2020. Σημαντικές πολιτικές κατευθύνσεις θα πρέπει να χαραχθούν από τώρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να δω ε, ποια είναι η αρχή της αλληλεγγύης, ε, της δαθικότητας θα μείνουν, δεν θα μείνουν νεκρό γράμμα, αλλά θα μεταφραστούν σε συγκεκριμένε δράσεις και πολιτικές. Αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να ε, ξεχνάμε την ε, θεμητή δυσπιστία και απομάκρυνση των πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή, στη μη στραφή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλού. θα πρέπει να περάσουμε από τις δυνατότητες της πράξης, από τις ενθουσιώδεις ε, δηλώσεις που θα γίνουν αύριο μεθαύριο στη Ρώμη, αυτή την εβδομάδα αλλος ιδιαιτέρως ε, της επαιτίου και μετά να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια για νέους κανονισμούς. Ε, το σχέδιο του, της συναδέλφου περιλαμβάνει πολλές, πολλές ενθαρρυντικές λαβές. Ε, από την θέση αυτή την ε, μακροοικονομική θα πρέπει να δούμε ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτική συνοχή και της ε, διακυβέρνησης της οικονομικής θα πρέπει να είναι δεμένη. Το περίφημο άρθρο 23 ε, της ε, παραπληρωματικότητας θα μπορέσει εδώ να βρει μια σωστή διατύπωση, τουλάχιστον ε, με πρωτοβουλίες να μην νερωθεί μετά και να μην παραλλαχθεί από τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Και αυτή η Επιτροπή, η ΡΕΤΖΙ, θα πρέπει να δώσει ένα σημαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα για να χαράξει το δρόμο προς το νέο κανονισμό. Εκεί όπου ρωτά, όπως στην παράγραφο 7 από την Κομισιόν, να δώσει μια αναπάντηση ε, και μία νέα προσαρμογή, νέο προγραμματισμό, που όμως θα είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περιφέρειας. Φυσικά, εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στα όσα συνέβησαν ε, το καλοκαίρι και το αθινόπερο υπό το φως των φρικτών ε, φυσικών καταστροφών του καλοκαιριού και του φθινοπόρου, να προβλέψουμε πιο, πιο ευέλικτο προγραμματισμό που θα σέβεται τα επιχειρησιακά προγράμματα θέματα των περιφερειών. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι όφελος. Τώρα, ε, όσον αφορά τους δείκτες για την κατανομή των πόρων, ε, όπως ε, λέει στην παράγραφο 15, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, και να βασιζόμαστε στις τρεις πυλώνες και δεν, που δεν είναι βέβαια τέλεια μεθοδολογία όμως το να τα όλα αυτά υπόψη και να προσπαθούμε να μετρήσουμε με ακόμα καλύτερα κριτήρια τη δυνατότητα μιας κοινωνίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μεμονωμένων πολιτών ας πούμε την πρόσβαση στο, στο υγειονομικό σύστημα την πρόσβαση σε στέγη να μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα ορίσουμε θεωρούμε πως είναι ε, απαραίτητο και να μας απασχολήσει. Τώρα, στις παραγράφους για τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουμε εκφραστεί διάφο... αρκετές φορές για το ΕΦΣΥ, για το ότι δεν είναι διαφανές και για το Omnibus υπάρχει κοκκίνδυνος να περάσουμε σε ένα απόλυτο πράσινο φως μεταφοράς των διευθυντικών ταμείων στο νέο σχέδιο Juncker. Ε, ελπίζω το κείμενο να μην αλλάξει και θέλω να το πω αυτό ε, σαφώς. Εάν δεχτούμε αυτού του είδους την κατεύθυνση και τη συνεργασία, όπως τις μεταρρυθμίσεις της διαρθωτικής του τότε να ξέρετε πως η πολιτική συνοχή μας θα ε, είναι πλέον νεκρή γιατί θα τις αφαιρέσουμε κάθε ουσία. Η πολιτική συνοχή δεν θα πρέπει να αποτελέσει το ε, σωσίβιο σωτηρίας για οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Να κλείσω με μια, μια ιδέα που έρχεται από πολλές ε, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι πολίτες περιμένουν μηνύματα για μετά το 2020, όπως την αφαίρεση των κονδυλίων των διευθυντικών ταμείων από το χρέος. Ελπίζουμε πως όλα αυτά θα μπουν στις ε, τροπολογίες και έτσι να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η εισήγηση ε, από την ε, ομάδα μας εδώ και από την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω τρία ακόμα ονόματα στον κατάλογο για τη συζήτηση. Υπάρχει άλλος κανείς, Βανίστελ Ρόι κυρία Μόλκοβα, ο κύριος και... Μάλιστα. Ωραία. Όλοι σας, όλοι σας. Σας βάζω στο λίστα. Μάλετιτς, κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές για τις εισηγήσεις τους. Είμαι ευτυχής που όλοι συμφωνούμε ότι η πολιτική συνοχής είναι μια βασική πολιτική, εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον <coughs> της Ευρώπης. Θέλουμε η Ευρώπη να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης, ε, ισχυρή και καινοτόμα, αλλά πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη πως η Ευρώπη είναι τόσο δυνατή όσο είναι το πιο αδύναμο κράτος μέλος της. Γι' αυτό και η πολιτική συνοχή είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί αφορά την αλληλεγγύη, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την βιώσιμη και την καινοτόμα ανανέωση. Σίγουρα η πολιτική συνοχής δεν είναι ευκολότερη, γιατί είναι μια πολιτική που θα έπρεπε εντόνως να είναι συντονισμένη με οριζόντιο και κάθετο τρόπο και, τα κράτη και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ένωσης. Και πιστεύω πως όλοι έχουμε κάποιο προβληματάκι με αυτό το καλό συντονισμό της πολιτικής συνοχής, γιατί κατά κάποιο τρόπο, ακόμα και στα κράτη-μέλη, αλλά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται χωριστή πολιτική. Θα έπρεπε λοιπόν στενά να συνδέεται με όλα, γιατί αφορά την απασχόληση, την αγορά εργασία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενέργεια, περιβάλλον, παιδεία, επιστήμες, τα πάντα καλύπτει. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι οι διάφορες ε, ε, γενικές διευθύνσεις δεν είναι τόσο καλά συντονισμένες και δεν συντονίζονται ούτε με την διεύθυνση που είναι αρμόδια, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική και μετά στα κράτη-μέλη επίσης τα Υπουργεία που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, κατά κάποιο τρόπο επίσης ε, χωρίζονται και ε, σαν να βρίσκονται σε παράλληλο κόσμο σε σχέση με τα υπόλοιπα Υπουργεία και αυτό η έλλειψη συντονισμού ε, μεταφράζεται σε έλλειψη αποτελεσμάτων και συνοχής. Ε, πρέπει να βρούμε τρόπο λοιπόν να συνεργαστούμε. Διότι η πολιτική συνοχής θα πει συνεργασία και συντονισμός. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, ε, είναι μια πολιτική αλληλεγγύης. Αν αυτό δεν το καταφέρουμε, ε, δεν θα έχουμε ούτε και αποτελέσματα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσεις για το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πιο συντονισμένα. Οριζόντιος συντονισμός και κάθετος συντονισμός. Και αυτό ε, ε, ε, σημαίνει εμπλοκή τοπικών, περιφερειακών, εθνικών αρχών, επιχειρηματιών. Όλα τα επίπεδα των, της κοινωνίας θα πρέπει να εμπλακούν εάν θέλουμε να χαρούμε τους καρπούς της πολιτικής συνοχής. Διότι ίδιοι οι πολίτες είναι αυτοί που θα επωφεληθούν περισσότερο. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το ενισχύσουμε στην έκθεση, το συγκεκριμένο σημείο και κάτι ακόμα είναι η ανάγκη η παράλληλη εργασία σε αυτή την περίοδο το 2017 και 2018 να εργαστούμε παράλληλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου αλλά και στο επίπεδο των κρατών μελών για την εφαρμογή του 2014-2020, πώς θα επιταχυνθεί δηλαδή η εφαρμογή πώς ε, θα δημιουργηθούν περισσότερες δυνατότητες ε, και θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία των project, αλλά ταυτόχρονα τώρα θα πρέπει άμεσα να εργαστούμε για την ε, κανονισμό τρομελοντικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για επιχειρησιακά προγράμματα το 2019. Θα είναι πολύ αργά. Το μάθημα αυτό το έχουμε διδαχτεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Να αρχίσουμε από τώρα να συζητάμε για το 2020 και να αρχίσουμε την εφαρμογή τους ήδη από το 2020, όχι το 2021. Ευχαριστώ πολύ. Νίλσον έχει ζητήσει το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. ξεκινώ λέγοντα ότι το προσχέδιο τη έκθεση που έχουμε μπροστά μα είναι μια καλή βάση συζήτηση. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι πώ μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Απλώ λέω ήδη από την αρχή ότι το κείμενο είναι εξαιρετικό. Σε τρία-τέσσερα σημεία όμω εγώ θα ήθελα να σταθώ και να προτείνω βελτιώσει. Πρώτα απ' όλα η απλοποίηση. Βεβαίως χρειάζεται, χρειάζονται προϋποθέσεις ε, και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την απλοποίηση, ωστόσο πρέπει να τονίσουμε και την ευθύνη των κρατών μελών. Ε, εμείς έχουμε αναλύσει την κατάσταση σε διάφορες σουηδικές περιφερειές, οποτεδήποτε διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με υπερβολικούς κανονισμούς και υπερβολική γραφειοκρατία και το αποτέλεσμα αυτή της ανάλυσης ήταν ότι το, η ευθύνη δεν βάρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν το κράτος μέλος, ήταν η γραφειοκρατία του κράτους μέλους που δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Άρα αυτό νομίζω θα πρέπει να φαίνεται πιο ξεκάθαρα στην έκθεση. Δεύτερο σημείο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Νομίζω ότι κάθε περιοχή χρειάζεται ένα σύστημα χρηματοδότησης, το οποίο θα βοηθά τις τοπικές επιχειρήσεις και τη συνεργασία μεταξύ τους. Από τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ε, προβλέπει χρηματοδότησης θα πρέπει να το κατευθύνουμε εκεί ακριβώ εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή στους συνεταιρισμούς, στις αγροτικές περιοχές, και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει Για, για, για τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα θα πρέπει να έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτο θέμα που θα ήθελα να αναδείξω και νομίζω ότι θα μπορούσε να ε, φάνει πιο ξεκάθαρα στη τελική έκθεση είναι ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά ταμεία και συχνά υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Το διαπιστώνουμε αυτό στη, στα διαφθορωτικά ταμεία όταν έχουμε ένα πρόγραμμα που αφορά μια περιφέρεια ε, που θα μπορούσε να υποβληθεί και σε περιφερειακό ταμείο ή σε διαφθορωτικό ταμείο. Πάντως, αναδεικνύοντας αυτά τα τρία ζητήματα, πιστεύω ότι το, το αρχικό που βάλει ο συγητής είναι ήδη πολύ καλό. Επόμενο ο ο κ. Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ την εισηγητρία το προσχέδιο εκθέση που έχει υποβάλει και για την ανταλλαγή απόψεων που κάνουμε. Κατά μία έννοια το σχέδιο αυτό της έκθεση. το έχουμε προετοιμάσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια με τις συζητήσει που κάνουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτή τη συζήτηση στην τελική έκθεση. Θα διοργανώσουμε τον Ιούνιο επίσης το φόρουμ για την συνοχή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις με ακόμα περισσότερους. Και ε, με χαρά διαπιστώνω ότι η συγκήτρια αξιοποίησε απόψεις που έχουν εκφραστεί στο παρελθόν. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά που είπαν ε, συνάδελφοι. Εγώ είμαι στα χέρια μου αυτό το έγγραφο που αναφέρεται στο μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ευρώπη και ερχόμαστε στα λόγια της κυρίας Μάλτσικ. Παρουσιάζονται ορισμένα σενάρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το βιβλιαράκι και το μόνο συμπέρασμα λογικό στο οποίο μπορεί να καταλήξει κανείς είναι ότι χρειάζεται συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να προχαρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άκουγα εχθέ τον κύριο Κατάινεν. Και ουσιαστικά αυτό μας έλεγε είναι ότι όλοι όλοι μαζί πιλοτάρουμε το αεροπλάνο. Ένα πρόβλημα έχουμε, μόνο ότι δεν βλέπουμε το αεροδρόμιο. και αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα συμμετάσχει και θα αγαπήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ένας πολίτης ε, ε, παρά μόνο εάν ε, του δοθεί, δεν του, α, παρά μόνο αν του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει. Δηλαδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό ή α, ασαφές η συνοχή, η πολιτική συνοχή είναι ο τελικός στόχος. Το βλέπουμε και στη συζήτηση για την κρίση. Ο κόσμος κατηγορεί τους τραπεζίτες και τώρα εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, πρέπει να βρείτε τη λύση. Το ερώτημα λοιπόν τελικά υπάρχει πραγματική συμμετοχή των πολιτών. Γιατί σε ορισμένες περιφέρειες βλέπουμε να ε, φεύγει ο πληθυσμό, να ερημώνουν εξαιτία τη εσωτερική μετανάστευση φεύγει ο κόσμο, πάει να εργαστεί στη Γερμανία για παράδειγμα. Και τελικά τι προτείνουμε σε αυτές τις περιοχές, να ερημώσουν άποψη μου είναι εναλλακτική, είναι να βελτιωθεί ή υπάρχει εναλλακτική. Ε, κατά την άποψή μου η εναλλακτική είναι να βελτιωθεί η περιφερειακή πολιτική ο δεύτερο πύλωνα της ΚΑΠ, η αξιοποίηση του στρατηγικού, του, του στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων. Αναφέρομαι στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, τι διαφορετικά δεν θα είχε νόημα, θα δίναμε, ε, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει για την ανάπτυξη τη περιφέρεια η ΚΑΠ. Θα λέγαμε ότι όλα τα χρήματα θα πάνε στον πρώτο πυλώνα, θα τα δώσουμε στου ε, γεωργού και τελείωσε. Ενώ μέσω του δεύτερου πυλώνα μπορούμε να προωθήσουμε και άλλου τύπου ε, ανάπτυξη, όπω για παράδειγμα ε, καινοτομία στι καλλιέργειε, τα ενεργειακά κτλ. Και χρειάζεται να βρούμε και έναν τρόπο επικοινωνία με του πολίτε. Πώ θα, θα, θα περάσουμε αυτό το, το μήνυμα ότι αντιποκρινόμαστε σε αυτά που θέλουν. Και να, μην, να εξηγήσουν στους πολίτες ότι, δεν, ότι και εκείνοι κατευθύνουν προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε. Ήμουν στο Άχιν το προηγούμενο στις Γερμανίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και πιο πριν στη Φραγκφούρτη και πιο πριν στο Βερολίνο και συνομιλούσαμε πολίτες, με έβρισκαν στον δρόμο πολίτες και μου έλεγαν μας αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, θέλουμε να συνεχίσουμε παρά τα προβλήματα. Άρα ε, πρέπει να αξιοποιήσουμε την ε, ευκαιρία που μας δίνουν τέτοιου τύπου συζητήσεις για να, καταλάβουν τι θέλουν, να καταλάβουμε τι θέλουν οι πολίτες. Και κάτι ακόμα. Για το ζήτημα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, συμφωνώ με τον συνάδελφο, δεν έχει νόημα να δίνουμε χρήματα έτσι ε, χωρίς κανέναν κανονισμό, χωρίς καμία προϋπόθεση και να τους λέμε ξοδεύστε τα. χρειάζεται να τηρούνται οι συμφωνίες ε, και αυτά που έχουν συμφωνήσει όσον αφορά την ε, δημοσιονομική ε, σταθερότητα και διακυβέρνηση. Για το συγκεκριμένο σημείο βεβαίως θα χρειαστεί να συνεργαστούμε περισσότερο με τη συνάδελφο για να καταγράψουμε στην έκθεση τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στην πράξη. Έχουμε κάποιες εμπειρίες από την Πορτογαλία και άλλες χώρες του Νότου, την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 δισεκατομμύρια διαθέσιμα στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, μέσω του ΕΦΣ. Και το ερώτημα είναι πώς θα τα εξοπλίσουμε αυτά. Προβλέπεται η χρηματοδότηση αυτή να αξιοποιηθεί 2018. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη φέρουμε πιο νωρίς. Ε, και επίσης γιατί δεν ανταμείβουμε εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν καταφέρει να επιτύχουν τους στόχους. Γιατί δεν αντιμείβουμε αυτούς που τα καταφέρνουν καλά. Δεν... Θα μιλήσω περισσότερο για συγκεκριμένες τροπολογία. Θα έρθω στο ζήτημα των συνεργειών, με το οποίο, στο οποίο βεβαίως όλοι συμφωνούμε και μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις περί της μεθοδολογίας και του συστήματος. Όμως, αν σκεφτούμε πόσο διαφορετικές είναι οι διάφορες περιοχές της Ευρώπης μεταξύ τους, στόχος θα έπρεπε να είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε μια περιφέρεια να βλέπει εκείνες που αποτελούν υπόδεγμα, που είναι πιο μπροστά, για να πάρει ιδέες. Και επίσης χρειάζεται να επιταχυνθεί η πολιτική μας για την συνοχή. για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Interreg. Πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη κατεύθυνση και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και υποδείγματα, πιλωτικά προγράμματα που να ε, λειτουργούν ως καλό παράδειγμα για τους άλλους. Πριν από δύο χρόνια είχα προετοιμάσει μια έκθεση για το ζήτημα της ε, βιομηχανίας και διαπίστωσε ότι υπάρχουν περιφέρειες στη Βουλγαρία, στη Σουηδία και αλλού όπου θα μπορούσαν να προοδεύσουν και να τα καταφέρουν στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν υποδείγματα, παραδείγματα, καλά παραδείγματα για να τονώσουμε την πολιτική συνοχής. παλιά συζητούσαμε για τις μεταλλαγές στον χώρο της βιομηχανίας. Έτσι το αντιμετωπίζαμε το ζήτημα της αλλαγής στη, στη βιομηχανία. Σήμερα ο όρος της μόδας είναι η βιομηχανία 4, 4-0, όπου πηγαίνουμε σε μια οικονομία όπου οι επικοινωνίες έχουν το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη σημασία. Πρωτοβουλίες σχετικές υπάρχουν σε διάφορα ε, μέρη της Ευρώπης. Και όπως είπε και η κυρία Μέλτεμπερκ, σε αυτόν τον τομέα δεν έχουμε επαρκή πολιτική επενδύσεων. δεν προσφέρεται το εύση γιατί το ρίσκο είναι υψηλό. Δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα μέσω του Horizon 2020. Άρα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ίσως συμπληρώνοντας μια τροπολογία για να αναφερθούμε συγκεκριμένα στο θέμα. Σας ευχαριστώ, κυρία Μόλκοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε πολλά από αυτά που ήθελα να πω υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί ε, καραδοκούν ε, και μηχανεύονται διάφορα οι εχθροί της συνοχής. Κάθε φορά που προετοιμάζουμε μια νέα πολιτική ή ε, μια νέα προγραμματική περίοδο επταετίας, θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα διάφορα δεδομένα και κάθε φορά πρέπει να τρέχουμε να πείθουμε τους πάντες ε, ε, ότι είναι σκόπιμη η περιφερειακή πολιτική, ότι παραμένουν περιφέρειες καθυστερημένες κάτω του 75% και χρειάζονται ενίσχυση. Τα ίδια ζήσαμε και το 2014. Ήταν οι φίλοι της συνοχής, αν θυμάστε τότε, στην Πρατισλάβα. Ε, συναντήθηκαν 14-15 κράτη-μέλη και ήταν παρόν και ο Μάρτιν Σούλτς ε, και ε, ήθελαν να σώσουν την πολιτική ε, συνοχή στον προϋπολογισμό ήδη από το 2014. Και τώρα τα ίδια ακούμε. Ε, πάλι διάφορες φωνές κατά της πολιτικής συνοχής και με διάφορα επιχειρήματα που ορισμένα ευσταθούν κιόλα. Και, και εμείς τους δίνουμε αυτά τα επιχειρήματα. Η Επίτροπος ήρθε στην Επιτροπή μας, δεν έμεινε πολύ ώρα, της έκανα μια ερώτηση, δεν μου την απάντησε. Και τι γίνεται με την επταετή αυτή προγραμματική περίοδο. Υπάρχουν χώρες που απορροφούν μόλις 3%, 3%, 3 της πολιτικής συνοχής. Τα γνωρίζω όλα αυτά. Ξέρω ότι τα προβλήματα ε, είναι και στα κράτη-μέλη, όπως είπε η κυρία Μάλετιτς, και μετά μην ερχόμαστε να εκπλησόμαστε που στον κανονισμό Omnibus έχουμε και τέτοιες προτάσεις ε, μεταφοράς πιστώσεων αλλού. Εχθές συζήτησα με τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών και προσπαθούσε να με πείσει ότι ε, δεν θα χαθούν οι πόροι, θα παραμείνουν στα κράτη-μέλη. Μια μικρή μεταφορά πιστώσεων κάνουμε. Ναι, ωραία. Και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές θα επενδύσουν ακριβώς στις πιο φτωχές περιφέρειες και εκείνες που θα έχουν περισσότερο ανάγκη. Γιατί η πιθανότητα τίνει στο μηδέν θα πρέπει να αγωνιστούμε για την πολιτική συνοχή και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει εδώ συνεργάτες και να ακούν αυτά που λέμε και τις παρατηρήσεις μας και να τις σημειώνουν. Επίσης, θα ήθελα να καλέσω την Προεδρία του Συμβουλίου να καταβάλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή, να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε στο μέλλον την πολιτική συνοχής. Γιατί πολύ συχνά ακούμε ότι ναι, ναι, αλλά δεν διαβιβάζονται αυτά αρμοδίως. Φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το σχέδιο Juncker και ε, δεν ε, μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ε, χρόνο έχουμε, αλλά να πιέσουμε και να ρωτήσουμε τις χώρες που απορροφούν μόλις το 3% γιατί δεν στέλνουν τα χρήματα στις περιφέρειες. Θα μπορούσα να σας δώσω παραδείγματα από τη δική μου χώρα. Αλλά χρειάζεται να ταρακονηθούν, να δοθεί μία προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν και ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες ε, που ε, πλήττονται ιδιαίτερα. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, και εγώ να ε, χαιρετήσω την έκθεση της κυρίας Βέσφαλ. Είναι πολύ χρήσιμη για την Επιτροπή μας και τα θέματα που θα μας απασχολήσουν αργότερα. Συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις που κάνετε, ιδιαίτερα την απλοποίηση, τα θέματα των χρηματοδοτικών μέσων ή ακόμα και ε, αυτά που προτείνεται για την πολιτική συνοχή να φτάνει σε όλες τις περιφέρειες. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω σε ένα τμήμα της έκθεσης, ιδιαίτερα στην παράγραφο 12, που ασχολείται με το θέμα της αναλογικότητας και της διαφοροποίησης. Ε, μέγα πρόβλημα ε, της πολυπλοκότητας απορρέει από τη λογική την ίδια. Ε, ότι θέλουν να εφαρμόζεται ομοιόμορφα και ενιαία η πολιτική αυτή ανεξαρτήτως χώρας, περιφέρειας, ποσού ή διοικητικής δομής. Ε, το κρατάω αυτό που αναφέρεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διαφοροποίηση και θα πρέπει ε, να είναι στο κέντρο κάθε προβληματισμού για τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Ήθελα να επιμείνω σε αυτό. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά μας και θα αποτελέσει ε, βάσει το έγγραφο της εκθεσής σας για μελλοντική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριος Μπόγοβιτς. Ευχαριστώ πολύ την συγκήτρια για την εξαιρετική πραγματικά έκθεση. Ε, νομίζω ότι περιλαμβάνει όλα τα κρίσιμα και σημαντικά σημεία. Έχει έρθει η ώρα να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή στην Επιτροπή μας. Ε, ε, γιατί είμαστε εμείς ακριβώς ε, ακρεφνείς υπέρμαχοι της πολιτικής συνοχής. Η πολιτική συνοχής είναι ορόσημο από τα σημαντικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις τέσσερις ελευθερίες είναι ένα βασικότατο στοιχείο ε, που πραγματικά ενώνει τις περιφέρειες. Θα πρέπει να σχεδιάζεται καλά και να εφαρμόζεται ακόμα καλύτερα. οι μεταρρυθμίσεις που είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής ε, συνοχής πρέπει να συνεχιστούν. Εμείς πρέπει να βοηθούμε τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένα κριτήρια και ενθαρρύνσεις. Ε, πολύ συχνά τα κριτήρια αυτά θεωρούνται εμπόδια και ακόμα καταγγελίες και παράπονα. Ε, δείχνουν όμως μια κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 η πολιτική αυτή συνόδευσε την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη νέα ε, προγραμματική περίοδο οι στόχοι έχουν αλλάξει. Διαπιστώνουμε δυσκολίες στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε σχέση με τους πόρους από το ε, ορίζοντα 2020 που έχουν απορροφηθεί μόνο το 5% ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, το 95% των κονδυλίων πήγαν στις παλιές λεγόμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη για να απορροφούν πραγματικά τα κονδύλια. Έχει μεγάλη σημασία ε, η πολιτική αυτή να αρχίσει το συντομότερο και το συντομότερο ε, να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη στη χάραξη, στην εκπόνηση της πολιτικής αυτής. Να ξέρουμε που οδεύουμε, αλλά και τα κράτη-μέλη από την αρχή για να αποφεύγουμε καταστάσεις τύπου απορρόφηση 3% μόνο. Από εκεί και πέρα η έκθεση τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε δυσκολίες. Δεν το αφισβητώ στα διάφορα κράτη-μέλη όπου παραμένουν οι διαφορές ανάμεσα στις περιοχές και τις αγροτικές υπαίθρου και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μεταναστεύσεις και μετακινήσεις από την υποανάπτυκτη νότιο-ανατολική περιφέρεια προς την βορειοδυτική. Μετά υπάρχουν διαφορές και στο εσωτερικό των κρατών μελών, οι πιέσει ε, μεταναστευτικές και προσφυγικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περασμένο Σαββατοκυριακό ε, πήγα στην Αλβανία Νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια προς τις χώρες αυτές που είναι εκτεθειμένες στη μεγαλύτερη πίεση για το μεταναστευτικό. Τα κράτη-μέλη και τα κράτη της συνοχής συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας, της πατρίδας μου, θα πάρουν 3, με 7 χιλιάδες ε, κατά στο μέλλον. Στα Δυτικά Βαλκάνια το αντίστοιχο ποσό ε, δεν υπερβαίνει τα 300 έως 700 ευρώ ε, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα χάσμα το οποίο θα επηρεάσει την πολιτική συνοχή αλλά και την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και το κόστος του Brexit που θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε και να βρούμε και περισσότερα χρήματα για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, κυρία Τόμασιτς. Thank you very um, Ευχαριστώ την θεία για το σχέδιο έκθεση. Συμφωνώ μαζί της ότι είναι καιρός να προετοιμάσουμε την πολιτική συνοχή για να μπορέσουμε να αρχίσουμε όντως στην αρχή του νέου προγράμματος. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες και την οικονομική και κοινωνική ε, συνοχή να προωθηθεί σε όλες τις περιφερειές της Ένωσης. Αυτό που δεν συμφωνώ ή μάλλον δεν στηρίζω την δράση που προτείνει η η συγκήτρια είναι να προτείνει δηλαδή μακροοικονομικούς όρους γιατί αυτό είναι μία από τις προστέμενες αξίες αυτής της πολιτικής. Επιπλέον, αν θέλουμε να έχουμε μια εξυγχρονισμένη πολιτική συνοχής, δεν λείπει εστιασμό στην λείπει μάλλον ο εστιασμό στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, πιστεύω πως ε, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στις στρατηγικές εφιούς ειδικευσής για να μπορέσουμε να έχουμε ε, συνδυασμό με δραστηριότητες οικονομικού τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να συμμετέχω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι μία από τις πιο σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Αν και συμφωνώ πλήρως πως όλες οι συζητήσεις ε, στην ε, Επιτροπή Ρέντζι μας προετοιμάζουν για αυτή την έκθεση όπου συγκεντρώνονται όλες οι θέσεις της Επιτροπής Ρέντζι για το επόμενο φόρουμ για τη συνοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της και να πω ότι συμφωνώ με τα βασικά μηνύματα που περιλαμβάνει αυτή όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες θέσεις ε, άλλες ε, δικές μου. Καταρχάς, συμφωνώ με τους συναδέλφους που υπογράμμισαν τη συσχέτιση μεταξύ μακροοικονομικών όρων και πολιτικής συνοχής, διότι ε, θεωρώ πως δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πολιτική συνοχής από την μακροοικονομική ανάπτυξη τον επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η πολιτική είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μελών. Στην ουσία λέει ότι αυτό είναι κομμάτι ολόκληρης της διαδικασίας της μακροοικονομικής ανάπτυξης. Οπότε το να διατηρήσουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στη μακροοικονομική ε, μακροοικονομικούς όρους και τη συνοχή είναι ένας τρόπος για να υπογραμμίσουμε το ρόλο της πολιτικής αυτής. Δεύτερον, στηρίζω το ρόλο των, δημοσιονομικών μέσων γιατί προσελκύουν ε, ιδιώτες επενδυτές και άλλους πόρους ε, της Ένωσης. Είναι σημαντικό να συμπληρώνονται τα δημοσιονομικά μέσα και πολιτικές. Αλλά δεν έχουμε, ε, συζητάμε συχνά τη συμπληρωματικότητα με το ΕΦΣΙ, αλλά όχι με την πολιτική γεωργίας και η ο συνδυασμό των πολιτικών αυτών είναι πολύ σημαντικό για κάποιε περιφέρειες και συμφωνώ με του συναδέλφου που λένε για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα σε αυτέ τι πολιτικέ. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να συνδέονται. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα γίνουν παραπληρωματικές και στα πώς θα συντονιστούν αυτές οι δύο πολιτικές. Να τονίσω και το εδαφική συνεργασία. Ε, προετοιμάσαμε μάλιστα και μια ειδική έκθεση και υπογραμμίσαμε την προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας, διασυνοριακή συνεργασία, όπως η συνεργασία για την οποία μιλά ο κύριος Μιλτεμπορκ που είναι μία από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής ως πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα στις περιφέρειες είτε μια ίδιας χώρας είτε και χωρών που είναι όμορες είτε και χωρών που δεν έχουν κάνει κοινά σύνορα. Θα έλεγα λοιπόν να συμπεριλάβουμε εδώ και την ειδίκευση και την καινοτομία γιατί ήδη έχει αποδειχτεί η προστιθέμενη αξία κατά την εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής. Και κάτι ακόμα που αναφέρεται κυρία Βέσβαλ, την ορατότητα της πολιτικής Πρέπει όχι μόνο να υπερασπιζόμαστε την πολιτική, αλλά να την καταστήσουμε πιο ορατή και πιο κοντινή στους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική η συζήτηση αυτή και θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Thank you κύριε Ιωάννη, για τις δικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα προλάβα να ε, καλύψω όλα τα θέματα που αναφέρθηκαν. Ξεκινώ λέγοντας ότι το προσχέδιο της έκθεσης ε, το θεωρούμε μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ως το 2020 και έρχεται σε μια ε, επίκαιρη χρονική στιγμή. Πιστεύω ότι η κυρία Βέσφαλ κατάφερε με τρόπο επικοδομητικό να συνοψίσει τη συζήτηση. Θα ήθελα να απαντήσω σε μία-δύο παρατηρήσεις που έκαναν μέλη του Κοινοβουλίου ξεκινώ με ένα από τα θέματα που ενδιαφέρει όλους μας, τα αγαπημένα μας, είναι το ζήτημα της απλοποίησης. Θα συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Νίλσεν, φαντάζομαι κανείς δεν εκπλήσεται από αυτό, ότι χρειάζεται συμμετοχή και των αρχών των εθνικών που παρακολουθούν τα προγράμματα για διάφορα ε, συγκεκριμένα ε, ζητήματα Όταν ακούμε ιστορίες από διάφορα κράτη-μέλη και διαπιστώνουμε ότι για το ίδιο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό κάποιος πρέπει να σε μια χώρα συμπληρώνει πέντε σελίδες αίτηση και σε άλλες 50 σελίδες αίτηση, ε, πρέπει να βρούμε μια λύση. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να συνομιλήσουν μεταξύ τους τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές αρχές για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες που έχουν ε, για την διαχείριση, στον τομέα της διαχείρισης των ε, ταμείων συνοχής. Θα ήθελα επίσης όμως να πω και να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ρεαλιστική και άρα να είναι ξεκάθαρο τι εννοούμε με τη λέξη απλοποίηση, γιατί υπάρχει η τάση συχνά να αναφερόμαστε στην απλοποίηση εννοώντα την απλοποίηση των διαδικασιών στο ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή στην περίπτωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μιλάμε για μια απλοποίηση η οποία θα κάνει τη δικιά μα δουλειά, τη δουλειά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο εύκολη. Το ζήτημα όμω θα ήταν και αυτό που θα βοηθήσει στην πραγματικότητα, ε, πώ μπορούμε να απλοποιήσουμε το πρόγραμμα ή την πολιτική για τι διαχειριστικέ αρχέ. Για το ζήτημα του αναπραγματισμού που ανέφερε ο κ. Φαν Μίλτεμπουργκ. Ε, και συμφωνώ και διαφωνώ Εγώ θεωρώ ότι ο αναπρογραμματισμός θα πρέπει να είναι πολύ εύκολος διαδικαστικά μιλώντας, δηλαδή από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση για αναπρογραμματισμό. Αυτό να ε, μπορεί να διεκπεριωθεί γρήγορα. Από την άλλη, και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Κιωφάν Μιλτέμπορκ, δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να ληφθεί αυτή η απόφαση. Γιατί θα πρέπει να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι εταίροι του προγράμματος να μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση για να αποφασιστεί αν είναι όντως η κατάλληλη στιγμή να γίνει ένας αναπρογραμματισμός. Θα συνόψιζα την κατάσταση λέγοντα ότι τα έχουμε καταφέρει, έχουμε καταφέρει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια διαδικασία η οποία είναι πολύ περίπλοκη. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ στο, σε ορισμένε παρατηρήσει που έγιναν για το πώ μπορούμε να ενθαρρύνουμε ε, την ε, συνεργασία μεταξύ περιφερειών. Είναι ξεκάθαρο ότι ο προπολογισμό, ο διαθέσιμο στο πλαίσιο του Interreg δεν είναι επαρκή. Και κάποια στιγμή μάλιστα θυμάμαι ότι το ποσοστό των, των προγραμμάτων που αποτύχαναν ήταν στις τάξεις του 90% και αυτό οδηγεί και σε ένα φαύλο κύκλο. Μετά δεν έχουμε αιτήσει σε αυτά τα προγράμματα. Στόχος λοιπόν θα ήταν να ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ περιφερειών στο πλαίσιο των περιφερειακών ταμείων. Γιατί όπως γνωρίζετε η το είπε και ο κύριος Φανίστελ Ρόι, ε, υπάρχουν ορισμένες περιφέρειες που είναι πιο μπροστά από τις άλλες. Υπάρχουν τέσσερις ε, συγκεκριμένες περιφέρειες οι οποίες προσπαθούν προσπάθησαν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να ε, στήσουν ένα πρόγραμμα διαπεριφερειακό και τελικά μόνο δύο συμμετείχαν. Επομένως δεν αξιοποιούνται πλήρως και όπως θα έπρεπε ε, όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν και όλη η ευελιξία που προβλέπεται στους διάφορους κανονισμούς. Και οποτεδήποτε διαπιστώνουμε τέτοιο τύπο αποτυχίες πρέπει να ξαναγυρνάμε και να εξετάζουμε τι δεν λειτουργήσε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί οι διάφορες αρχές δεν αξιοποίησαν αυτά τα προγράμματα. Όσον αφορά την απορρόφηση γενικά, Είναι ένα θέμα το οποίο ανέφεραν και μέλη της Επιτροπής σας. Οι απόψεις διήστανται όσον αφορά την απορρόφηση. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να ε, μετρήσουμε την απορρόφηση. Εάν εξετάσουμε την, την απορρόφηση στο επίπεδο των προγραμμάτων ανά κράτος μέλος, πολλά κράτη-μέλη τα καταφέρνουν καλά. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, το 80% ε, της χρηματοδότησης που της αναλογεί έχει ήδη αποδοθεί σε προγράμματα και ε, τελευταία νέα ε, μας λένε ότι η Ουγγαρία μέχρι το τέλος της χρονιάς θα καταφέρει το 100%. Όσον αφορά λοιπόν την απόδοση κονδυλίων σε προγράμματα τα πράγματα λειτουργούν. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ χειρότερα ε, όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Για πολλά κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πλευρά τη ε, στις συζητήσεις που έχει στις επιτροπές παρακολούθησης με τα κράτη-μέλη. Δεν αρκεί να κοιτάει κανείς μόνο το εάν τα κονδύλια έφτασαν στους δικαιούχους. Το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί έντονα στις Βρυξέλλες είναι ότι οι πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί δεν υλοποιούνται ακριβώς επειδή δεν υλοποιούνται τα προγράμματα, επειδή δεν προχωράει η απορρόφηση. Οποιαδήποτε βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα αυτό θα μας βοηθήσει γιατί είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε και, και στα κράτη-μέλη. Έρχομαι τώρα στο περιεχόμενο της ίδιας της έκθεσης. Ομαδοποιώντας τα διάφορα θέματα. Ε, όπως θα το φαντάζεστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με όλα αυτά τα παρατηρήσει που διαβάζουμε στην έκθεση για την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων αυτών, την σημασία της εταιρική σχέσης, την συμμετοχή και οριοσοντίως και καθέτως των διαφέρων εταίρων. Νομίζω. Αυτό είναι ξεκάθαρο ξεκάθαρο πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής. Δεν είναι απλό να υλοποιεί κανεί την πολιτική συνοχή με αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν πιο εύκολο διαδικαστικά μιλώντα να υπάρχει ένας, ένα κεντρικό σύστημα συντονισμού. Αλλά εάν κάναμε κάτι τέτοιο δεν θα είχαμε αποτελέσματα στην πράξη στις, στις διάφορες Όσον αφορά την αρχιτεκτονική. Συμφωνούμε με πολλά από τα στοιχεία της έκθεσης. Για παράδειγμα, τη σημασία που αποδίδεται στην ευελιξία, στην εκ των προτέρων αρισιμότητα. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, εντός της Επιτροπής του Κοινοβουλίου ε, διστάμενες απόψεις όσον αφορά το κατά πόσο είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε την μακροοικονομική ερεσιμότητα. Ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει η πολιτική συνοχή στα κράτη-μέλη θα ήταν να αξιοποιηθεί για να ενθαρρύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Να λειτουργήσει ως κίνητρο δηλαδή η πολιτική συνοχή έτσι ώστε τα διάφορα κράτη-μέλη, οι διάφορε περιφέρειε των κρατών μελών να κινηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή να κάνουν τι δαπάνε του αποτελεσματικότερε μακροπρόθεσμα. όσον αφορά τους κύριους τομείς πολιτικής, συμφωνούμε με αυτό που αναδεικνύει και η έκθεση ότι η καινοτομία έχει μεγάλη σημασία. Αυτό χρειάζεται να το φροντίζουμε και σε επίπεδο πολιτικής γενικό και σε επίπεδο υλοποίησης στην κάθε ε, περιφέρεια και στο κάθε έργο. Το ζήτημα είναι πώς καταφέρνει κανείς να καλύπτει ε, συνολικά τους διάφορους τομείς πολιτικής. Δεν θα μπορούσε κανείς ρεαλιστικά να περιμένει ότι με ένα έργο ε, θα καλύπτει όλους τους τομείς πολιτικής, με κάθε ένα έργο ξεχωριστά, αλλά αν κοιτάξουμε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από την συνοχή συνολικά, ε, θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε σίγουροι ότι καλύψαμε τα πάντα. Ε, τελικά αυτό σχετίζεται και εξαρτάται από τι διάφορε συζητήσει και τι διάφορε διαπραγματεύσει που κάνουμε με του εκπροσώπου των περιφερειών για το ποιε είναι οι ανάγκε του και ποιε τομεί πολιτική θα πρέπει να καλύπτουν. Ένα τομέα στον οποίο υπολοιπόμαστε είναι η αντιμετώπιση των συναπιών τη παγκοσμιοποίηση και των τεχνολογικών αλλαγών. Θα έλεγε κανεί ότι ο λόγο ύπαρξη τη πολιτική συνοχή ήταν να αντιμετωπίσει ακριβώ αυτά τα θέματα. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία ελοποιείται η πολιτική συνοχή δεν είναι επαρκή. Θα έπρεπε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ε, αλλαγές, αυτές τις προκλήσεις πιο γρήγορα από ό,τι το καταφέρνουμε σήμερα για να προσαρμοζόμαστε πιο γρήγορα. Τέλος, συμφωνώ με την ε, σημασία που δίνεται στο ζήτημα της δημοσιοποίησης, της ε, προβολής. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε και ο κ. Φανίστηλ Ρόι στην παρέμβασή του. Η Επιτροπή προετοιμάζει μια ανακοίνωση για το πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα σε αυτό το τομέα. έτσι ώστε αυτά που γίνονται στην, μέσω της πολιτικής συνοχής να προβάλλονται σε όλα τα επίπεδα. Κλείνω λέγοντας ότι σας ευχαριστώ για αυτή τη ε, συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα συμμετάσχουμε φυσικά και στο Φόρουμ Συνοχής Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, η συγγετρία. Ήρθε η ώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, δεν θέλω να μακρηγορήσω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η συζήτησή μας έδειξε πόσο σημαντικό είναι για μας το θέμα, κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο, ότι ανησυχούμε για το μέλλον. Πώς να το διατυπώσω τώρα. Ανησυχούμε μήπως ε, μας επιφυλάσσει το μέλλον μια διαφορετική πολιτική συνοχής που δεν την επιθυμούμε εμείς. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος ε, που θέλουμε να εστιάσουμε το κέντρο βάρους. Θυμίζω ότι είναι έκθεση πρωτοβουλίας και πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε γιατί είμαστε περιορισμένοι στο μήκος της έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, για τις προτάσεις σας, την πληθώρα προτάσεων και τροπολογιών φαντάζομαι θα κάνετε πολλές. Απλώς το είπα από την αρχή θα υπάρξουν κάποια πράγματα που δεν τα βλέπουμε με το ίδιο μάτι. Γι' αυτό είναι διαφορετικά τα κόμματά μας και οι πολιτικές ομάδες και δεν είμαστε όλοι στην ίδια. Τελικά όμως θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, διότι όπως καταλαβαίνουμε είναι η αρχή και μόνο της συζήτησης για το πώς θα διαμορφωθεί μια μελλοντική πολιτική συνοχής. Και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε αυτό το ενακτήριο λάκτισμα ακολουθούν δύο πολιτικά επίπεδα, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα πρέπει να τα αναγκάσουμε να ασχοληθούν και πάλι με την πολιτική συνοχής και να τη συνεχίσουν με ε, διαφορετική μορφή, βελτιωμένη, όχι με λιγότερα χρήματα, αλλά περισσότερα. Και αυτό είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε και σκληρή μάλιστα και θα πρέπει να είμαστε καλά οπλισμένοι. αυτό προηγουμένως το είπα, όχι επειδή φοβάμαι μήπως έχουμε διαφορετικές γνώμες και τροπολογίες και μήπως διαφωνήσει κανείς μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι για να είμαστε ισχυροί θα πρέπει να έχουμε μια στεναρή φωνή για την πολιτική συνοχή και όσο γίνεται πιο ενωμένη. Να δείξουμε την κατεύθυνση από εκεί και πέρα ε, βελτιώσεις ε, σε λεπτομέρειες θα γίνουν και αλλού, θα υπάρξουν και άλλες εκθέσεις όχι στην παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμείς να δώσουμε τη μεγάλη κατεύθυνση προς τα που θέλουμε να βαδίσουμε εμείς ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ως Κοινοβούλιο και θα αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια για να υπερασπιστούμε την πολιτική συνοχή μας απέναντι σε όλους τους εχθρούς και τις αντιστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για τις απολογίες σας που σίγουρα θα είναι πολύ άριθμες και το θέμα θα είναι συναρπαστικό και στις συζητήσεις των σχεδόν θα τα δούμε αυτά τα θέματα και τελικά θα έχουμε καλή έκθεση, έτσι λέει η πείρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θυμίσω την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 30 ε, Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Και προχωρούμε στην επόμενη έκθεσή μας για σήμερα το πρωί. Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχή. Είναι η έκθεση τη κυρίας Ρούζα Τόμασιτς. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχει ήδη γίνει για την έκθεση αυτή. Πέρσι, τον Νοέμβριο μάλιστα, το 16 έγινε αυτό. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης και θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Προτείνω να ρίσουμε μια προθεσμία για τις τροπολογίες. Παρασκευή 24 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Τόμασης για να μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της Παρακαλώ τους συναδελφούς, κάντε λίγη ησυχία. Κυρία Τόμασίτς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η τεχνική αρρωγή είτε είναι πρωτοβουλία της ε, Επιτροπή των Κρατών Μελών είναι απαραίτητη σε όλες τις φάσεις εξέλιξης των προγραμμάτων της συνοχής και είμαι ευτυχής που αναγνωρίζεται η σημασία αυτής της έκθεσης. Υπάρχει ακόμα χώρος για βελτίωση του ελέγχου και, της και την αξιοποίηση της τεχνικής αρρωγής παρά το γεγονός ότι η προγραμματική περίοδος 2014-2020 κυρίω έχει εστιάσει στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ευρεία στρατηγική για την τεχνική αρρωγή που θα περιλαμβάνει όλες τις ε, κύριες διοικητικές ε, δομές που εργάζονται για τα ε, διορθωτικά προγράμματα ώστε να αποφευθεί η επικάλυψη, ενώ θα να προωθηθεί η συνεργασία και η συμπληρωματικότητα έχει αναπτυχθεί έτσι ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων για την αυτοεκτίμηση, αυτοαξιολόγηση, καθώς και συμβάσεις για τον έλεγχο των πολιτών. Έχουν δημιουργηθεί ευέλικτα και προσαρμόσιμα ε, μέσα τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις διάφορες οργανωτικές δομές των κρατών μελών. Ε, στόχος είναι να υπάρξει η ε, τεχνική αρρωγή ώστε να μπορέσουν να φτάσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και να αυξηθεί η διαφάνεια και η ευθύνη στα στις δημόσιες δομές. Να αυξηθεί επίσης η εμπιστοσύνη των δημοσίων οργάνων στους δημόσιους διαγωνισμούς, να αυξηθούν αυξηθεί η αξιοπιστία των ε, ε, ε, συμμετεχόντων και να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή στην αγορά. Η τεχνική αρρωγή φτάνει στα 13,7 δις στο πλαίσιο των διευθυντικών ταμείων. Αυτός είναι ένας παράγοντας αλλαγής, όμως η συμβολή του μπορεί να εκφραστεί μόνο στο μέλλον όταν οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν ολοκληρωθεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο σχεδιασμός, συντονισμός και η διαφάνεια να είναι εγγυημένες σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής. Είναι σημαντικό να είναι εγγυημένος ο ρόλος των τεχνικών μεταρρυθμίσεων για τις διαρθρωτικές πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ε, νομιμότητα. Το τεχνικό τμήμα θα πρέπει να μην δαπανάται από Ε, μάλλον να δαπανάτε ε, παράλληλα με την εθνική χρηματοδότηση που δεν θα πρέπει να την αντικαταστήσει. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη εξήγηση για τις πολιτικές συνοχής. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας κάθε προτινόμενου προγράμματος είναι και το επίπεδο ευαισθητοποίησης. Οι πιθανοί υποψήφοι θα πρέπει να έχουν όλες τις πληροφορίες για τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την άποψη της τεχνικής αρρωγής. Καλό λοιπόν τα κρατημέλη να ενημερώνουν καλύτερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της τεχνικής αρρωγής και για τα αποτελέσματα. Περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ορατότητα της τεχνικής αρρωγής, ώστε να ε, μπορέσουν να ε, γίνουν και οι κατάλληλες ε, ενέργειες, αλλά επίσης ε, να ε, υπάρξουν και οι βάσεις δεδομένων που προβλέπονται. Μετά το 2019 ε, θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες για να συμπεριλάβουμε και τα συμπεράσματα Ε, του προγράμματος αυτού. Δυστυχώς πολλά κράτη-μέλη στην τεχνική αρρωγή χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο για να ε, καταρτιστούν οι εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών δομών. Όμως δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα όλοι αυτοί να εκφράσουν τις απόψεις τους και άρα η κατάρτιση δεν είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες αυτές. Τώρα είμαι ευτυχής για τη συνεργασία για, με τους ε, σκιώδη εισηγητέ και είμαι πεπισμένη ότι η κοινή μα προσπάθεια θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητα για την τεχνική αρρωγή. Ευχαριστώ. Και θα μιλήσει εξ τη κύριε Σπυράκη από το ΕΛΚ, ε, ο κύριο Βανίστερ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της εισηγήτριας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται τις δυνατότητες που έχουμε από την πολιτική συνοχή και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Η κυρία Τόμαζιτς ε, ε, επισήμανε τα πιο σωστά σημεία. Έχει έρθει η ώρα της διαφάνειας και της λογοδοσίας για το πώς ε, δίνεται αυτή η τεχνική αρρωγή και πώς αξιοποιούνται τα κονδύλια. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Κάθε φορά εκπλησόμαστε όταν ε, ως Περιφερειακή Επιτροπή πηγαίνουμε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε τις διαπραγματεύσεις και μετά βλέπουμε ότι 140 εκατομμύρια τα πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για ποιο λόγο, διότι δεν απορροφήθηκαν. Μα πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι πάει στραβά. Φτιάχνουμε ένα κατάστημα και βγάζουμε ε, έτσι, όλα τα εμπορεύματα και παίρνουν απόλυτα, γιατί δεν έρχεται πελάτης. Hello, ακούει κανείς. Ε, πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Είναι πολλά τα λεφτά και μπαίνουν αναπορόφητα. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη τέτοιες εκθέσεις μετά. Και η κυρία Σπυράκη λοιπόν υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να μελετήσουμε την κατάσταση σε μεγαλύτερο βάθος και στην Task Force για την Ελλάδα, για παράδειγμα, την οποία αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας, υπάρχουν κάποια πράγματα που πήγαν εξαιρετικά καλά και άλλα που είναι εμπόδια και πρέπει να υπερπηδηθούν ή να αρθούν για τις μεταρρυθμίσεις σε αυτή την προσέγγιση αναχώρα έτσι, που έχουμε προγράμματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους για να αποφύγουμε και επικαλύψεις υπάρχει ας πούμε μια συμβουλευτική, ένα συμβουλευτικό κόμβος, ένα νέο μέσο για τις επενδύσεις, ε, ένα νέο εργαλείο που τον Απρίλιο ε, θεσπίστηκε στην Ολομέλεια. Και κάνουμε επενδυτικές προσπάθειες και εμείς έτσι ώστε να ε, πιάνουν τόπο τα χρήματα, η προσέγγιση να είναι ε, στοχευμένη με εστίαση στο αποτέλεσμα και μπορεί να χρειάζονται και κάποιοι δείκτες επιδόσεων για να μετράμε τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής και να δαπανούμε τα χρήματα αποτελεσματικά. Σύμφωνο με την εισηγήτρια λοιπόν και με την κυρία Σπυράκη για την έκθεσή σας. Και έχω και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Σκοτσολίνο. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Έχω τρία ερωτήματα, ε, τρία θέματα μάλλον, επί των οποίων ίσως θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Το πρώτο είναι το θέμα των τοπικών αρχών. Πώς η τεχνική αρρωγή στηρίζει την εμπειρία που διενεργούν. Έχουμε σημαντική εμπειρία στο εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά τώρα ξεκινά ε, ένα πρόγραμμα τεχνικής αρρωγής για τις ε, αστικές περιοχές. Εκεί δεν έχουμε ακόμα αρκετή εμπειρία. Δεύτερο είναι πώς η τεχνική αρρωγή, κυρίως αυτή που έχουμε λάβει σε ορισμένα κράτη, αλλάζει την ποιότητα των ε, διοικητικών παροχών. Δηλαδή, στην ουσία γεννιέται μια νέα κουλτούρα στη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων, ιδιαίτερα για τις περιφέρειες όπου ε, δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν τα, τα κοινοτικά ταμεία. Η τεχνική αρρωγή είναι μία πρώιμη και πνευματική εργασία που μπαίνει μέσα σε πλαίσιο ενός μηχανισμού ή μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη εμπειρία που τροποποιεί επίσης τη διοικητική δομή στην καθημερινότητα της διεκπαιρέωσης των ε, δημοσίων ε, υποχρεώσεων. Κάτι ακόμα που θα πρέπει επίσης να τονίσουμε είναι το σημείο 16 όπου τονίζεται το θέμα της τεχνικής αρρωγής που και περισσότερο προσανατολίζεται στους παραλήπτες και στην ποιότητα των project. Και εδώ πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, γιατί συχνά η τεχνική αρρωγή είναι τεχνική αρρωγή για τους θεσμούς και δεν είναι τόσο για αυτούς που στη συνέχεια πρέπει συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που εμείς τους διαθέτουμε. Πρόκειται για εταιρείε, πρόκειται για πανεπιστήμια, πρόκειται για μεμονωμένους δικαιούχους των διευθυντικών ταμείων. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτού πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο και να πούμε και κάποια περισσότερα λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος κοιόδης εισηγητής είμαι εγώ η ίδια. Θα κάνω μια μικρή παρέμβαση και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδελφούς. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση για την τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα να καλωσορίσω ότι ε, βασική βασική ε, θέση της εισηγήτριας ότι πρόκειται για έναν οριζόντιο και γενικό τομέα. Χρειάζεται να αξιολογήσουμε την προστεθέμενη αξία αυτής της τεχνικής βοήθειας. Επίσης θα ήθελα να ε, επισημάνω τα εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, ε, θα πρέπει να προετοιμάσει μια αξιολόγηση εξ για την τεχνική βοήθεια και για την στις περιπτώσεις όπου η τεχνική βοήθεια ε, γίνεται με κεντρική διαχείριση και, και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μεικτή διαχείριση. Γιατί εστιάζουμε περισσότερο στις περιπτώσεις της τεχνικής βοήθειας από τα κράτη-μέλη μεταξύ κρατών μελών και δεν δίνουμε την ίδια σημασία όταν η βοήθεια παρέχεται από την Επιτροπή κεντρικά. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ε, εφαρμογή του κανονισμού για την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις, τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν χρειάζεται να, συνεργαστεί το, ε- να, να συνδυαστεί το ΕΦΣΥ με άλλα ε, προγράμματα χρηματοδοτικά. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη λειτουργία του επενδυτικού κόμβου και το ένα. και το, η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να την εξετάσουμε από την πλευρά των δικαιούχων, δηλαδή των διαχειριστικών αρχών και το πώς αυτές μπορούν να αξιοποιούν τα ταμεία συνοχής με βάση το θεματολόγιο που έχουμε επιλέξει είναι, για τις αστικές περιοχές είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνική βοήθεια θα συνεισφέρει στην πολιτική μας για τις αστικές περιοχές. Πρέπει να βελτιωθεί επίσης η συνεκτικότητα της πολιτικής συνοχής με τις πολιτικές που προωθούμε μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ένα επίσης σημαντικός τομέας στον οποίο πρέπει να εργαστούμε είναι η βελτίωση της προβολής της πολιτικής συνοχής έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ε, από πού ήρθαν τα χρήματα, τι καταφέραμε με αυτά και πώς βοήθησε η τεχνική βοήθεια. Η τεχνική βοήθεια μπορεί να συνεισφέρει και σε αυτόν τον τομέα και φαντάζομαι θα το συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Σε ευχαριστώ κύριε Τόμασιτς, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες στην έκθεσή σας. Επόμενος σκιώδης, μάλλον η κυρία Ντεμάτο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ την συνάδελφο Ε, το θέμα της τεχνικής αρρωγής και ε, της, ε, των διοικητικών δυνατοτήτων είναι πολύ σημαντικό και ε, γι' αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη και γενικά στις νομοδοτήσεις. Η τεχνική αρρωγή θα έπρεπε να έχει το στόχο να, βοηθεί, να βοηθάει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα διάφορα προγράμματα και project που χρηματοδοτεί η Κομισιόν. Αυτή η βοήθεια οικονομικού τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία ε, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και ε, αυτοέλεγχο. Πολύ συγκεκριμένε προτάσεις γίνονται, όπως ε, έχουμε διαπιστώσει, οι δυσκολίες έχουν οι τοπικές αρχές για να έχουν συγκεκριμένο και ειδικευμένο προσωπικό σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτό είναι σημαντικό γιατί εμποδίζει όχι μόνο τις δυνατότητες των δημοσίων εργών να χρησιμοποιήσουν σωστά τα διευθυντικά ταμεία, αλλά και γιατί συχνά ιδιώτες και συμβουλευτικέ εταιρείε είναι αυτέ που βοηθούν τι διοικητικές δομέ, πολύ συχνά οδηγώντα σε σπατάλη, σε σπατάλη των δημοσίων χρημάτων. Τον Οκτώβριο του 2015, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, από μια δημοσιογραφική έρευνα ενός ε, εβδομαδιαίου ε, Ιταλικού περιοδικού, δύο συμβουλευτικέ εταιρείε φάνηκε ότι η Brian ε, Cooper και η Ernest Young 32 και 42 εκατομμύρια ευρώ ε, κέρδισαν από συμβουλευτικές ε, δραστηριότητες για την Νότια Ιταλία. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή, είτε για, καλύτερα, ναι, ή για να καταρτιστεί καλύτερα ο δημόσιος τομέας, αλλά αυτό κυρίως αφορά το θέματα ε, ε, των περιφερειών και των κρατών μελών, είτε για να προσληφθεί κατάλληλο προσωπικό στο δημόσιο τομέα. Επίσης είναι σημαντικό και κρίσιμο ε, να δούμε ποια είναι τα πραγματικά ωφέλη για όσον αφορά τη στήριξη των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων που τελικά ε, οδηγούνται σε άλλου σκοπούς. Συμφωνούμε αντίθετα στο να επιστηθεί η προσοχή στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Διοντολογία για την εταιρική σχέση, έτσι ώστε οι εταίροι να μπορέσουν να βοηθηθούν, να ενισχύσουν τις δικές τους θεσμικέ δυνατότητες για να μπορέσουν να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν τα προγράμματα. Τέλο, είναι απαραίτητο να γίνει μια ανάλυση όπου η τεχνική αρρωγή θα πρέπει να είναι ένα συν μέσα σε κάθε πρόγραμμα. Μια αξιολόγηση για το ποια από τις δύο λειτουργίες είχε περισσότερα αποτελέσματα και επέφερε βελτιώσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση, ώστε να μπορέσουμε έτσι να οδηγηθούμε ε, σε καλύτερο, να μάλλον να τα λάβουμε υπόψη στην επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού και των κατευθυντηρίων γραμμών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νίλσεν, είστε επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντική η τεχνική αρρωγή ώστε να ε, αξιοποιηθεί πλήρως το κάθε project, ε, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα προγράμματα. Δεν είναι πάντοτε δυνατό να γίνει όμω να χρησιμοποιήσουμε τεχνική αρρωγή, γιατί πρέπει να ανατρέξουμε στι εθνικέ αρχέ. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει διευκόλυνση τη συνεργασία για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε αυτή την κατευθύνση σωστή, αλλά να είμαστε πιο κάθετοι και πιο συγκεκριμένοι στι παρεμβάσει μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής μας, όχι. Παρακαλώ τον Επίτροπο, συγγνώμη, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπόιμανς, τμήματάρχης ε, στη DG Regio για ε, θέματα ανταγωνιστικότητας. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα μέσα καλύτερα στο μέλλον Στην τεχνική βοήθεια στην περίοδο 14 20 καλούμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα τη βοήθεια αυτή. Στο παρελθόν δίναμε ένα ποσό κατά αποκοπή για την τεχνική βοήθεια και δεν ασχολείται πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δαπάνη των χρημάτων αυτών. Καλούμε τα κράτη-μέλη λοιπόν να είναι πιο στοχευμένα και να βελτιώσουν τα στρεβλά των προηγουμένων περίοδων. Τα περισσότερα πηγαίνουν σε ανθρωπίνους πόρους, σε κόστος προσωπικού. Για μισθούς, πριμ και πόνους. Θα πρέπει έτσι να το κάνουμε πιο σωστά και να μείνουμε και να, μάλλον, να επιβλέψουμε καλύτερα τους ενδιάμεσους προϋπολογισμούς ε, και κονδύλια που χρησιμεύουν στα μικρά προγράμματα πολύ. Επίσης, ε, ε, ελέγχουμε τις μη πληρούμενες, τους μη πληρούμενους εξάντε όρους, καθώς και ελέγχουμε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα για να μπορέσουμε να, να ε, ε, ε, με βάση τα νέα μέτρα κατά των απατών. Εάν πετύχαμε όλα όσα θέλαμε να πετύχουμε, όχι βέβαια, αλλά θέλουμε να μπορέσουν να δαπανηθούν τα χρήματα με πιο αποτελεσματικό ακόμα τρόπο. Μπορούν να υπάρξουν και άλλες βελτιώσεις. Πρόκειται για ένα έγγραφο αυτό εδώ το οποίο μπορεί πολύ καλά να ενταχθεί στη συζήτηση. Κάποιο κομμάτι της τεχνικής αρρωγής επίσης θα μπορούσε να προκαταβληθεί και να χρησιμοποιηθεί ε, πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν τις δυνατότητες να ε, ε, χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια αυτή και στη διαδικασία της επιλογής και της εφαρμογής. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην να δούμε μάλλον πώς, ποια θα είναι η εξέλιξη και όχι να γίνει μια ολόκληρη επανάσταση ή ανατροπή του συστήματος, απλώς να χρησιμοποιηθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο και πιο ενισχυμένο. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον ε, για να μπορέσουμε να, πάω, να, να χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες δυνατότητες στο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε την πλήρη ολοκλήρωση και την πιο αποτελεσματική χρήση της τεχνικής βοήθειας από όλα τα ταμεία. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια στρατηγική για όλα τα ταμεία και με ε, συνδυασμό και εκ των υστέρων αξιολόγηση για το πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνική βοήθεια και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συνδιαχείριση σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Είναι καλό να εξάγουμε τα διδάγματά μας για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια αυτά. Έγιναν διάφορα σχόλια για να προσθεθούν και άλλοι δικαιούχοι. Ε, θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και την διοικητική δυνατότητα και ικανότητα των δικαιούχων και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια στο βαθμό που είναι πάντα ε, στοχευμένη για τους δικαιούχους που απορροφούν περισσότερα ε, περιφερειακά κονδύλια, διαφθορτικά ταμεία που είναι βασικά οι αρχές της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Μας έγινε και μια άμεση ερώτηση για την υποαπορρόφηση σε κεντρικό επίπεδο της τεχνικής βοήθειας. Καταρχάς, Πρέπει να σας πω ότι στη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο, τουλάχιστον για αυτή την προγραμματική περίοδο, έχουμε στρατηγική για τη χρήση τεχνικής βοήθειας. Είναι 8-9 οι προτεραιότητες, δηλαδή επικεντρωνόμαστε σε τομείς ε, κλειδιά που είναι σημαντική ε, αστική ανάπτυξη, ε, δυνατότητα διοικητική κλπ. Κάτι άλλο που πρέπει και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βελτιωθεί η τεχνική βοήθεια σε κεντρικό επίπεδο είναι να αναζητούμε συστημικές λύσεις και συστηματικές αντί για πρωτοβουλίες ad hoc. Ας πούμε να δίνουμε τα χρήματα σε οργανώσεις όπως είναι το Jasper, σε διάφορα συστήματα ομοτήμων peer-to-peer, αντί να έχουμε ατομικές, εξατομικευμένες και αποσπασματικές λύσεις, ένα γενικότερο σύστημα που μπορούν να κινητοποιηθούν περισσότερα κονδύλια και να αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια, 142,9 εκατομμύρια δόθηκαν στο, στο πρόγραμμα ε, αναδιάρθρωσης ε, της ε, διορθωτικής πολιτικής. Δεν θα έλεγα ότι χάθηκαν τα χρήματα για τη συνοχή. Μιλάμε για επενδύσεις, κρατικές προμήθειες, κρατικές ενισχύσεις, εξυγχρονισμό υποδομών. Όλα αυτά έχουν όφελος έμεσο ή άμεσο από τους δικαιούχους των υπόλοιπων ταμείων. Αυτά προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόμασιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, θα, θα μακρηγορήσω κι εγώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι προτάσει του, για τι παρατηρήσει του. και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε επικοδομητικά όπω και σε αυτήν την ε, συζήτηση. Νομίζω θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή τελική έκθεση. Η πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Εδώ θα κλείσουμε την, ε, το πρωινό μέρο τη συνεδρίασή μα. Ε, η απογευματινή συνεδρίαση είναι στι 3 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επισκεφτούμε την εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Αντιπρόεδρος Ταγιάννη για τον εορτασμό της 60ης επαιτίου της συνθήκης της Ρώμης. Σας ευχαριστώ και καλό απόγευμα.